Τώρα έχουμε σε κοινή συζήτηση την έκθεση της κυρίας Σταρκεβιτσούτε σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές στην κοινότητα και την έκθεση John Purvis για τη δραστηριότητα Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Σταρκεβιτσούτε για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε. Σήμερα όπου η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως βρίσκεται σε κρίση είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις ε, οικονομικές δομές και να αναπτύξουμε την εσωτερική αγορά. Η εσωτερική αγορά είναι πολύ κατακαιρματισμένη, ιδίως όσον αφορά τις ε, ε, υπηρεσίες και θα πρέπει να δημιουργηθούν κοινέ δομές για τις διασυνοριακές πληρωμές. Το έγγραφο αυτό έχει μία ιστορία, διότι όταν ε, ε, ε, καταρτήσει και το ευρώ είχε διευκρινιστεί ότι οι διασυνοριακές πληρωμές και τα τέλη που που τα ε, επακολουθούν θα αναφέρονται ε, μέσω μίας ειδικής προτάσεως κανονισμού 2560 ε, και αυτή αναφέρεται στις διασυνοριακές πληρωμές τόσο εντός μίας χώρας όσο και ε, διασυνοριακά. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε να επιτύχουμε μια μεγαλύτερη, έναν μεγαλύτερο ανταγωνισμό εις ε, τις διασυνοριακές πληρωμές αλλά βλέπουμε ότι όταν μεταφέρει κανείς 100 ευρώ πριν ισχύσει ο κανονισμός πληρώναμε 24 ε, ευρώ ενώ τώρα το ποσό συρρυκνώθηκε σε 2,5 ευρώ και η πρόταση η νομοθετική πρόταση αποβλέπει ε, στην επαλήθευση της εφαρμογής του κανονισμού 2560 για να διευρύνει την εφαρμογή της διότι η εφαρμογή τώρα ε, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις περισσότερους τομείς και ε, αναφέρομενος στον κανονισμό αυτό θα μπορέσουμε να αλλάξουμε το τοπίο πληρωμών στην Ευρώπη ε, και αυτό βέβαια περιλαμβάνει διάφορες διατυπώσεις. Ο κανονισμός αυτός προβλέπει ότι όταν δεν υπάρχει σύμβαση μεταξύ ε, των δύο μελών ε, στην διασυνοριακή πληρωμή θα έπρεπε εφόσον πρόκειται για διασυνοριακές ε, πληρωμές να μην ε, ξεπερνά το επίπεδο τα 0,08 ευρώ και τα κράτη αυτά θα πρέπει να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους κατά τρόπον ώστε να καταρτήσουν τις αρχές οι οποίες θα πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους στα διάφορα κράτη-μέλη και ε, θα εντοπίσουν τα ασθενή στιμία ε, καταρτίζοντας κριτήρια που θα ελέγχουν αυτές τις διαδικασίες. Ένα άλλο έγγραφο το οποίο προτείνεται σε αυτό το έγγραφο είναι ε, η κατάργηση ε, ορισμένων ε, πληροφοριών που πρέπει να δίδουν οι τράπεζες ορισμένων κρατών αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί διότι και πρέπει να πω ότι δυστυχώς σε αυτό το σημείο δεν έχουμε συμφωνήσει με το Συμβούλιο και τα στατιστικά στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε δεν έχουν ακόμη καταρτιστεί και δεν έχουμε καθόλου στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριος για τέσσερα λεπτά. Uh, Η οδηγία αυτή ανταποκρίνεται στη μεγάλη ανάγκη του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ηλεκτρονικού χρήματος καθώς και στην ανάγκη να υπάρχει ένα σαφέ νομοθετικό πλαίσιο με στόχο να διευκολύνει τη χρήση του ηλεκτρονικού χρήματος ε, για ηλεκτρονικούς ε, λογαριασμούς, πληρωμή ε, τηλεφωνικών καρτών, κάποιων δώρο επιταγών κτλ. Επίσης όμως ορίζεται και η νομισματική αστυνομία ε, αξία και ορίζονται και ορισμένες ε, συναλλαγματικές ε, μετατροπές, πιστοτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, καλύπτει πληρωμές για μικρά χρηματικά ποσά συνήθως, σε επιχειρήσεις άλλες εκτός του χρήστη, κάποιες άλλες προπληρωμένες κάρτες, τηλεφωνικές και άλλες. Αλλά και σε περίπτωση που δεν χρειάζεται να έχει κάποιος λογαριασμό στην τράπεζα. Πριν από 8 χρόνια, ένας, ε, ο Μπέντζαμιν Κέρ στο άρθρο ηλεκτρονικό χρήμα έλεγε ότι σύντομα θα έρθει η μέρα του ηλεκτρονικού χρήματος. Δυστυχώς η πρόβλεψη ήταν και υπεραισιόδοξη αλλά και πρόημη για την Ευρώπη τουλάχιστον. Το ηλεκτρονικό χρήμα ακόμη δεν έχει δώσει τα αποτελέσματα και τα ωφέλη τα οποία αναμενόταν να έχει ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001 εγκρίθηκε η πρώτη σχετική οδηγία και αυτό ίσως ε, λόγω των αρχικών ε, κεφαλαιοκών απαιτήσεων και άλλων περιορισμών σε ό,τι αφορά το κόστος και υπάρχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματο από το ένα κράτο στο άλλο. Στην Τσεχική Δημοκρατία έχουμε πάνω από 40 παραδείγματο χάρη. EMI, δηλαδή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, ενώ δύο σημαντικές ε, χώρες, Γερμανία και Γαλλία, έχουν 12 μόνο και μάλιστα στην Γερμανία δύο ε, ιδρύματα τέτοια δεν θέλουν να εγκατασταθούν στη Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των σημαντικών ε, νομικών διαφορών που υπάρχουν. Τον Αύγουστο του 2007, δηλαδή πριν από δύο χρόνια, μόνο το ένα δις ευρώ ήταν ηλεκτρονικό χρήμα. Το ηλεκτρονικό χρήμα λοιπόν ακόμη έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι ότου γίνει μια σοβαρή εναλλακτική λύση αντί των μετρητών. Παρά τους περιορισμούς ε, έχουμε ακόμη προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσει νέες καινοτόμες και ασφαλίσει για το χρήστη υπηρεσίες ε, πληρωμών είναι αυτή η οδηγία να βοηθήσει την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες και να επιτρέψει τον ομαλό ανταγωνισμό μεταξύ των φόρων. Και οι μικροί πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στην αγορά καθώς θα μειωθεί από ένα εκατομμύριο ε, στα 350.000 ευρώ το κεφάλαιο που πρέπει να διαθέσει κανείς στην αρχή, το αρχικό κεφάλαιο. Βέβαια εμείς θα προτιμούσαμε ε, ένα χαμηλότερο ποσό. Επίσης ε, μπορούν να διευρυνθούν οι χώροι πληρωμών ο πελάτης μπορεί να πληρώνει πλέον πρέπει χάρη το εισιτήριο του μετρό με μια κάρτα, να αγοράσει τον καφέ του, να αγοράσει ένα μπουκέτο λουλούδια στα κιόσκια των σταθμών όπως γίνεται στο Χονγκ Κόνγκ με πολύ μεγάλη επιτυχία ήδη από τώρα. Έχουμε διατρέξει την νομοθετική διαδικασία έτσι λίγο γρήγορα για να εγκριθεί στην πρώτη ανάγνωση και πριν τις ευρωεκλογέ να εγκριθεί αυτή η οδηγία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, ακόμη και τη Μέλανη συγκεκριμένα, αλλά και τους σκιώδεις εισηγητές, επιτέλας ρεύα, τις υπηρεσίες της Κομισιόν, την Τσεχική Προεδρία και τον Τόμα Τρίνχον και την ομάδα του κυρίως για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε όλοι αυτοί. Βέβαια δεν έχει επιτύχει κανένα από εμά όλα όσα επιθυμούσε στην αρχή, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και πραγματικά θα ήθελα να ζητήσω την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο αυτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πίτροπε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πάνω απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ταχύτητα του Κοινοβουλίου στην εξέταση αυτών των δύο σημαντικών χαρτοφυλακίων. Και θέλω να ευχαριστήσω γι' αυτό και τους συζητητές και την Πρόεδρο Περβάνος Περές που συνέβαλαν με αποφασιστικό τρόπο στην ταχύτητα των εργασιών. Σήμερα λείπουν μόνο δύο μήνες από την ημερομηνία που τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν αυτή την οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Αυτά τα δύο μέτρα μαζί με την τομέα των πληρωμών που θα παράγει τα σωστά προϊόντα είναι σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς των πληρωμών. Τέτοια μέτρα μαζί με την οδηγία θα συμπληρώσουν την νομική βάση που είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε σαφήνια βεβαιότητα και σταθερότητα της αγοράς. Οι διαπραγματεύσεις που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες μας επέτρεψαν να πετύχουμε τάχιστα συνένεση όσον αφορά τα δύο αυτά χαρτοφυλάκια. Όσον αφορά τον κανονισμό που αναθεωρείται για τις συνολικέ πληρωμές, χαίρομαι που ανακοινώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την τροπολογία που προτάθηκε που ήταν καρπό συμβιβασμού. Τη δέχεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαίρεται ιδιαίτερως για τη συμπερίληψη στην αρχική της πρόταση άρθρων που θέτουν πλαίσιο για το θέμα της, δια... της πολυμερούς διατραπεζικής επιτροπής για τις, για τις συναλλαγές άμεσης χρέωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα για ε, την χρήση των ευρωπαϊκών, του στήματος αυτού από τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες. Αυτοί οι κανόνες θα δώσουν στον τομέα των πληρωμών τρία χρόνια για να προτείνει ο τομέας σε ένα εμπορικό μακροπρόθεσμο μοντέλο για την αυτόματη χρέωση σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την οπτική γωνία του συμβιβασμού είναι διαθέσιμη να αντικαταστήσει την κατάργηση ανεφόρων αυτών των υποχρεώσεων με μια ρήτρα επανεξέτασης όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Όσον αφορά την οδηγία για το ηλεκτρονικό χρήμα, την αναφερμένη οδηγία, πρόκειται περί νομοθεσίας άκρος φιλόδοξης που θα δώσει δεύτερη δυνατότητα ε, για τους φορείς να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό χρήμα. Θέλει να δώσει οδηγία στην αγορά ένα νομικό πλαίσιο και πλαίσιο συνετής διαχείρισης που θα είναι σαφές και ισορροπημένο, εξαλείφοντας άχρηστα εμπόδια, δυσανάλογα υπερβολικά όσον αφορά την είσοδο στην αγορά και κάνοντας πια ενδιαφέρουσα την δραστηριότητα ε, χρήσεως ε, ηλεκτρονικού χρήματο. Η οδηγία θα πρέπει να ευνοήσει πραγματικό και αποτελεσματικό ανταγωνισμό μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ταυτόχρονα όμω να εγγυάται ισότιμε συνθήκε για όλου του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών και να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Οι επιτευθέντες συμβιβασμοί πετυχαίνουν άριστη ισορροπία προστατεύοντας τους στόχους μας, τους αρχικούς και ταυτόχρονα ανταποκρινόμενοι στις θεμητές προσδοκίες και ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των συζητήσεων και θέτησης των μέτρων. Υποστηρίζουμε λοιπόν πλήρως αυτή την πρόταση για τους προναφερθέντε λόγους και σας ευχαριστώ. Εν ονόμα της Επιτροπής, Νομικής ο κ. Σακαλάς έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Νομική Επιτροπή στηρίζει την πρόταση αυτή σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές στην κοινότητα. Ε, ζητούμε καταρχήν να αντικατασταθεί ο ισχύων κανονισμός, δεύτερον να προωθήσουμε την προστασία του καταναλωτού και να δοθεί ε, το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για ένα αποτελεσματικό σύστημα πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτον ε, να μπορέσει να προωθηθεί το θέμα αυτό στην Ευρώπη. Η Επιτροπή μας μετέδωσε την ε, γνωμοδότησή της στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεσμάτων και αναφέρθηκε εις ε, τις διατυπώσεις που συνεπάγονται οι διασυνοριακές ε, πληρωμές για να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματα που τίθενται από αυτή την πρόταση. Πρέπει ε, να τονίσουμε ότι η αναλογικότητα και η επικουρικότητα πρέπει να ισχύσει και στις διασυνοριακές πληρωμές σύμφωνα με το άρθρο 95.1 της συνθήκης θα χρειαστεί να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση σε όλη την κοινότητα, να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι σε όλα τα κράτη-μέλη για να υπάρχει νομική βεβαιότητα και να μπορέσουν όλοι να είναι ικανοποιημένοι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι ομιλητές εν ονόματι των ομάδων καταρχήν ο κύριος, κύριος Γαρσία μαρισκάλου για, του ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα σχολιάσω μόνο τον κανονισμό για τις ε, διασυναριακές απληρωμές και την έκθεση της κυρίας ε, Σταρκεβιτσιούτε. Ο κανονισμός, όπως εξηγείται πολύ καλά στην έκθεση, ανταποκρίνεται στις ανάγκες οι οποίες εννοούνται ω ε, συνέπεια της εισαγωγής του ευρώ και θεσπίζει μια σχετικά σαφή αρχή θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι όροι για τις εθνικές και για τις διασυναριακές πληρωμές που είναι ένας ε, κανόνας κοινή λογικής στην εσωτερική αγορά αλλά ο οποίος ε, δεν είχε ε, τηρηθεί πριν από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Ξεκίνησε λοιπόν με το ευρώ και σιγά σιγά ο νέος χώρος πληρωμών σε ευρώ. Με το πέρασμα του χρόνου αυτός ο κανονισμός πλέον έχει απαρχαιωθεί και θα πρέπει τώρα να αναθεωρηθεί για να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών αλλά και στην οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τρεις στόχους έχει θέσει. Ε, πρώτα απ' όλα να συμπεριληφθεί στο πλαίσιο του κανονισμού ε, η διασυνοριακές ε, πληρωμές, εξοδικαστική επίλυση επίσης προβλημάτων που μπορούν να προέρχονται από την εφαρμογή του κανονισμού και τρίτον, ελάφρυνση, μετρίαση των ε, υποχρεώσεων στατιστικών πληροφοριών για το σωσίγιο πληρωμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί εν γέννη με το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, έχει ζητήσει τρεις σημαντικές τροποποίησεις. Διευκρίνηση των νομικών προϋποθέσεων και ορισμών που θα σπίζει ο κανονισμός Δεύτερον, συντονισμό ε, για τα κράτη-μέλη και προειδοποίηση ε, προς αυτά για να εφαρμόσουν καλύτερα τον κανονισμό από ό,τι στο παρελθόν. Ε, και τρίτον, μια επίκληση σε συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο ήταν η υποχρέωση για στατιστική ενημέρωση στον τομέα του ισοζυγίου των πληρωμών που ευτυχώς επιλήθηκε με συμφωνία των διαφόρων θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό και είμαι πλήρως ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα το οποίο έχει επιτευχθεί. Ευχαριστώ. Για σοσιαλιστές η κυρία Μπερέζ έχει το λόγο για δίλεπτον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τοποθετηθώ επί της εκθέσεως του κυρίου Τζον Πέρδης όσον αφορά το ηλεκτρονικό χρήμα. Καταρχάς πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε γιατί είναι λιγότερο εκπληγμένο εδώ το ηλεκτρικό χρήμα από ότι στο Χονγκ Κονγκ. Σίγουρα διότι οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν τις τραπεζικές τους κάρτες με μεγάλη ευκολία. Οι ανησυχίε αυτού του Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αφορούσαν δύο τομείς. Πρώτα απ' όλα τα θέματα της εποπτείας είναι στα χείλη όλων και δεν θέλαμε απλώς να πιεστούμε από τα λόμπι των Ιδρυμάτων Εκτονικού Χρήματος και δεν θέλαμε να απορριθμίσουμε λόγω της πίεσης την εποπτεία τους. Γι' αυτό μέρημα του Κοινοβουλίου ήταν αυτά τα Ιδρύματα που διαθέτουν ηλεκτρονικό χρήμα και το διαχειρίζονται να μπορέσουν πραγματικά να ελέγχονται. Και πετύχαμε κάποια χέγγια εκεί και χαίρομαι. Παρομοίως, θέλαμε να λάβουμε υπόψη τα συμφέροντα των πολιτών και εκείνων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό χρήμα. Κυρίως όταν θέλουν να διακόψουν τη σύμβασή τους. Για να μην τους επιβάλλουν τα ιδρύματα που χειρίζονται αυτό το χρήμα περιορισμούς και τέλη που θεωρούν υπερβολικά. Σε αυτό το πνεύμα υποστηρίξαμε αυτή την πρόταση. Θέλαμε να διευκολύνουμε τη ζωή των πολιτών μέσω της χρήσης του ηλεκτρονικού χρήματος. Αλλά αυτό δεν θέλαμε να οδηγεί σε παρεκκλήσεις, κυρίως όσον αφορά την εποπτεία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Για φιλευθέρους η κυρία Μπάεβα έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αναφέρομαι στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αποβλέπει στην αντικατάσταση του ισχύοντος κανονισμού ε, και αναφέρεται στην ολοκληρωμένη αγορά πληρωμών. Ε, αποβλέπουμε στο να ε, βελτιώσουμε την προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτού και να παρακολουθούμε τις στατιστικές. Στο άρθρο 5 του κανονισμού και στο άρθρο 12 όπου αναφέρεται η ρήτρα να θεωρήσεις καταλήξαμε σε συμβιβαστική λύση όπως βλέπουμε ε, στην έκθεση της κυρίας Σταρκεβιτσούτε και η Βουλγαρία συμφωνεί με την άποψη αυτή. Ε, θέλουμε να ε, υπάρξει μία βελτίωση των στατιστικών στοιχείων και εμείς είμαστε υπέρ της καταργήσεως των υποχρεώσεων ρυθμίσεως των τελών ε, για μεταβιβάσεις ε, κάτω των 50.000 ευρώ. Επίσης εμείς πιστεύουμε ότι ε, δεν θα πρέπει να μειωθεί η ποιότητα των στοιχείων που αναφέρονται στο ισοζύγιο πληρωμών και επιπλέον στο σύστημα για τις άμεσες πληρωμές. Ευχαριστώ. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ο κύριος Κράς δεν είναι εδώ, ούτε ο κύριος Λούινγκρεν, ούτε ο κύριος Γκοζές. Δεν ζητά κανείς ε, ε, σύμφωνα με τη διαδικασία Catch οπότε κύριε Επίτροπε αν θέλετε μπορείτε να απαντήσετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Για ακόμη φορά θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου για τον τρόπο με τον οποίο το Κοινοβούλιο χειρίστηκε αυτά τα δύο θέματα. Αυτό σημαίνει ότι ο νέος κανονισμός όσον αφορά τις συνορικές πληρωμές θα τεθεί σε ισχύ όπως προβλεπόταν την 1η Νοεμβρίου ενεστώτος έτους. Η αγορά του ηλεκτρονικού χρήματος θα έχει δεύτερη δυνατότητα έτσι για να αναπτυχθεί. Παράλληλα, η οδηγία όσον αφορά τι υπηρεσίε πληρωμών και οι διάφορες νομοθετικές πράξεις δημιουργήσουν το κατάλληλο σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο, γενικό πλαίσιο για την κοινοτική αγορά των πληρωμών και θα ανοίξει ο δρόμος ούτω ώστε η ευρωπαϊκό τομέα των πληρωμών να μπορέσει να αναπτυχθεί πλήρω και να δημιουργηθεί νέο χώρο πληρωμών σε ευρώ. Έτσι οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα εκμεταλλευτούν μια αγορά πληρωμών που θα είναι ολοκληρωμένη, αποτελεσματική, κυρίως όσον αφορά το κόστος και υψής της ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί λοιπόν και με ιδιαίτερη χαρά ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το μήνυμα ε, τη ε, υποχρέωση δέσμευση του Κοινοβουλίου να υποστηρίξει όλα αυτά τα μέτρα για το ηλεκτρονικό χρήμα και τις ηλεκτρονικέ πληρωμέ. Καλώ λέει Πρόεδρος. Πρόεδρο. Ο κύριο Λούντγκρεν απουσιάζει δεν ήταν εκεί και ήρθε τώρα. Θα του δώσω λοιπόν εκτάκτος μετά τον Επίτροπο. Όταν σας κάλεσα κύριε δεν ήσασταν εδώ, αλλά έχετε το λόγο τώρα. Για δύο λεπτά και μόνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, καλοσύνη σας. Ε, το ηλεκτρονικό χρήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διασυνοριακά είναι κάτι που αποτελεί σαφή πρόοδο και είναι ένα σημαντικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να βελτιώσει έτσι την εσωτερική αγορά προωθώντας τη χρήση αυτού του ηλεκτρονικού χρήματος. Δράτω με τις ευκαιρίες να υπενθυμίσω αυτά τα οποία συζητούμε. Περί τίνος πρόκειται. Όταν εισαγάγαμε το ευρώ για κάποιες χώρες, για σημαντικό αριθμό χωρών στην Ευρώπη, είχαμε βασιστεί στην ανάλυση που είχε διεξαχθεί ε, σχετικά με την αξία της νομισματικής ένωσης. Μπορούμε να μειώσουμε με τη σωστή προσέγγιση το κόστος των πληρωμών μέσω νομισματικής ένωσης. Αυτό σκεφτήκαμε. Ποιο είναι το τίμημα της νομισματικής ένωσης. Πιο ασταθείς οικονομίες. Ε, βλέπουμε την ανεργία που αυξάνεται. Είναι προβληματικό για τις χώρες να διατηρήσουν το ισοζύγιο πληρωμών τους. Το βλέπουμε τώρα χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα δεν τα πάνε καλά. Να σημειώσουμε λοιπόν εδώ ότι τα θύματα είναι εκείνα που υποτίθεται θα κέρδιζαν από τη μείωση του κόστους μέσω του ενιαίου νομίσματος. Η πρόοδος δεν επιτυχάνεται και έτσι ο σκοπός δεν επιτυχάνεται δεν επετεύχθη η πρόοδο στο ενοποιημένο σύστημα πληρωμών. Ελπίζουμε να φτάσουμε στην κατάσταση όπου το κόστο θα αναμεληταίο γιατί ε, οι πληρωμέ θα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και θα έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα το οποίο θα εγγυάται αστάθεια αν δεν πετύχουμε τους στόχου μας. Το είπα και προηγουμένως. Και βλέπουμε να συμβαίνει τώρα. Σκεφτείτε το λοιπόν, πρέπει να ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση. Πολύ καλά. Θα ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Σταρκεβιτσιούτη για δύο λεπτά. E, Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι το κείμενο εφαρμογής είναι το αποτέλεσμα μιας ενός συμβιβασμού μετά από μακριές διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω τους συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεργασία όπως επίσης και τους συναδέλφους που με βοήθησαν από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Και όπως είπε ο κύριος Λούντγκρεν, αυτή η νέα διάταξη θα βελτιώσει το σύστημα ΣΕΠΑ διότι θα υπάρχει καλύτερη ε, δυνατότητα χρήσεως του ευρώ. Η χώρα μου δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ αλλά χαίρομαι διότι αυτή η διάταξη θα μπορέσει να ισχύσει ακόμη και αν τα κράτη-μέλη ε, ε, δέχονται πληρωμές σε ευρώ και τα ε, μετατρέπουν στο εθνικό τους νόμισμα όπως το δικό μας. Ε, θα ισχύσει δηλαδή το σύστημα αυτό ε, για ε, εσωτερικές πληρωμές σε ευρώ και διασυνοριακές πληρωμές σε εθνικό νόμισμα. Θα χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτή η αρχή της διασυνοριακής διακπεραίωσης ακόμη και για το χώρο ο οποίος δεν ανήκει στη ζώνη του ευρώ. Η εφαρμογή αυτής της νομοθετικής διατάξεως επιτρέπει να εξυγχρονιστεί ο τραπεζικός τομέας διότι ο τραπεζικός τομέας εντός τριών ετών θα πρέπει να καταρτήσει ένα νέο πρότυπο το οποίο θα είναι πιο αποτελεσματικό διότι πολλές φορές μιλάμε για δαιμονοποίηση, για καινοτομία και πιστεύω ότι ακριβώς αυτή η διάταξη θα επιτρέψει κάτι να εξυγχωριστεί. Θα δώσω τώρα στον κύριο Πέρβη το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, η κυρία Περές ανέφερε κάποιες ανησυχίες στο τομέα της εποπτείας και πρέπει να πω ότι εμείς έχουμε επιμείνει στην οδηγία και στη σχετική έκθεση ότι τα ηλεκτρονικά ε, κονδύλα δεν αποτελούν καταθέσεις και δεν Πρέπει ε, να υπάρχει πίστοση σε αυτά. Οι βασικές κεφαλικές απαιτήσει έχουν μειωθεί για το αρχικό κεφάλαιο, δηλαδή σε 350.000. Εμείς θα, είχαμε, θα προτιμούσαμε 200.000, το ίδιο κεφάλαιο 2%, ε, εμείς θα θέλαμε 1,6%. Τέλος πάντων, με το 20% αυτό της ευελιξίας πάνω κάτω, τα πιο φιλελεύθερα μέρη μπορούν να φτάσουν στο 1,6% και στα συντηρητικά στο 2,4%. Δεν είναι ιδανικό, αλλά ε, υπάρχει αυτή η προοπτική. Υπάρχει ακόμα άνηση κανόνες παιχνιδιού, παρότι εμείς έχουμε ζητήσει τη διασφάλιση ε, κάποιων ε, διαδικασιών και κυρίως αυτό που ανέφερε η κυρία Μπερές θα πρέπει να υπάρχει επίσης ένα όριο και για εθνικούς παρόχους στα 5 εκατομμύρια ευρώ που δεν θα πρέπει να είναι 2 εκατομμύρια. Ένα προσεκτικό βήμα προς τα εμπρός, όχι τέλειο, έτσι είναι και κάθε συμβιβασμός. Σίγουρα θα πρέπει σε 3-4 χρόνια να επανεξεταστεί ο κανονισμός, αλλά ελπίζω να έχουν πει μέχρι τότε στην αγορά περισσότεροι υπάροχοι, να ζητούν και οι χρήστες περισσότερες επιλογές, ε, να υπάρχουν περισσότεροι ρυθμιστές, η κυρία Μπερέσια, η ΕΚΤ και όλοι οι άλλοι να έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για μια φιλική προς το χρήστη υπηρεσία που δεν θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή οικονομία και εμείς στην Ευρώπη να μπορούμε τελικά να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που προσφέρει το ηλεκτρονικό χρήμα. Σα ευχαριστώ. τέλο τη Στην ημερήσια διάταξη έχουμε τώρα την έκθεση Snell για υγειονομικού κανόνε σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Δίνω αμέσω το λόγο στον εισηγητή μα για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία